people here, so I καλώς ήρθατε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Γυναικών και ανάπτυξη. Πρόκειται για το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκή Ένωσης 2016-2020 για την ε, ισότητα των δύο φύλων. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν την παρουσίαση των ε, υπηρεσιών ε, εκπόνησης ερευνών. Είμαστε εδώ, όπως είπαμε, και από τις δύο επιτροπές και εγώ συμπροεδρεύω εδώ μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, την κυρία Λίντα Μακάβαν. Όπως ξέρετε, είναι μια σημαντική υπόθεση, σημαντικός φάκελος και για τις δύο επιτροπές μας που θέλουν να προωθήσουν την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων ως μια βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις πολιτικές και όλες τις δράσεις της. Αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα σε ένα κοινό εργαστήριο που έλαβε χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου και ακολούθησε μετά και ανταλλαγή απόψεων από κοινού μεταξύ μας στις 10 Οκτωβρίου. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε την δόκτωρα Ισαμπέλα Ιωαννίδες που είναι από την μονάδα για τις ex post αξιολόγησης του EPRS που θα μας παρουσιάσει την ε, μελέτη και την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος ε, δράσης ακριβώς για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Έχετε 15 20 λεπτά κυρία Ιαννίδης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ήταν μεγάλη μου χαρά να εκπονήσω αυτή την ε, έκθεση ε, για τις Επιτροπές ΕΝΤΕΒΕ και ΦΕΜ για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μάλλον θα γνωρίζετε ήδη ότι η μονάδα μας ε, για την εκ αξιολόγηση σε τακτική βάση εκπονεί τέτοιε εκθέσεις. Η συγκεκριμένη έκθεση αυτή έχει τρεις στόχους να εξετάσει την κατάσταση όσον αφορά τα επιτεύγματα. Ε, η τεχνολογία ε, δεν φαίνεται να λειτουργεί. Holding it in the right direction makes a difference. Ναι, αν το κρατάω σωστά, ε, λειτουργεί. Τρεις στόχους έχουμε λοιπόν, να εξετάσουμε την κατάσταση όσον αφορά τα επιτεύγματα του ΓΑΠ2, του νέου σχεδίου δράσης που θα συζητήσουμε σήμερα, τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής και να εντοπίσουμε πιθανές δυσκολίες ή ασυνέπειες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής του σχεδίου αυτού. Δεύτερος στόχος είναι να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε το πλαίσιο του ΓΑΠ, διότι εφαρμόζεται μόλις και ένα χρόνο ε, αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο δεν θα αναφερθώ πολύ στην παρουσίασή μου. Υπάρχει όμως τμήμα στην έκθεση που εξετάζει τα ε, συμπεράσματα που βγάλαμε από το σχέδιο δράσης 1 ε, καθώς και συγκριτικά, συγκρίσιμα αποτελέσματα από άλλα προγράμματα. όπου εξετάζεται ο ρόλος του φύλου. Και τρίτον, τρίτος στόχος είναι να εξάγουμε συμπεράσματα και να εντοπίσουμε ευκαιρίες για δράση στον τομέα αυτών. Κατά την εκπόνηση της έκθεσής μου, δύο παράγοντες επηρέασαν την επιλογή μεθοδολογίας. Καταρχάς, ε, το χρονικό διάστημα αξιολόγησης, μόλις ένα έτος δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι είχαμε ε, περιορισμένη διαθεσιμότητα ε, άμεσων δεδομένων και δεν είχαμε αρκετή απόσταση από τα γεγονότα. Κατά την εξέταση λοιπόν της πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θεώρησα ότι ήδη μιλάμε για ε, επιτυχή ε, ε, προγράμματα. Οι μέθοδοι λοιπόν που χρησιμοποίησαμε ήταν καταρχάς αξιολόγησης, αξιολογήσεις από ε, ομάδες προβληματισμού, think tanks, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους παράγοντες, ε, εκθέσεις τους χρησιμοποίησα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα από την Eurostat, τον OSA και ε, την ε, βάση δεδομένων της UNDP και είχα την ε, δυνατότητα να συνομιλήσω με διάφορες ομάδες προβληματισμού, με κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. και να πάρω στοιχεία από διάφορες εκδηλώσεις που είχαν οργανωθεί εδώ στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω πόσο σαφής είναι αυτή η διαφάνεια. Χρησιμοποίησα όμως τον δείκτη ανισότητας των δύο φύλων και έχω κατατάξει τα στοιχεία ανάλογα με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τις ε, διάφορες περιφέρειες για τα ε, οικονομικά μέσα που διαθέτει. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα το οποίο θα πρέπει να καλύψουμε. και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η δουλειά που γίνεται. Όσον αφορά τα συμπεράσματά μου, μέρος των επιτευμάτων συμπεριλαμβάνουν την ε, κατανόηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης ε, των ε, γυναικών. Αυτό συνάδει με τα βασικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, το στρατηγικό σχέδιο για την ισότητα 2016 2019. Έχουμε προχωρήσει πέρα από τα GAP 1, διότι ενώ είχαμε προσέγγιση σε τρία τμήματα, τώρα έχουμε ε, διευρύνει τις δράσεις ε, σε, σε, σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος των ανδρών ως παράγοντες ε, στην ε, διασφάλιση της ισότητας ε, των δύο φύλων. Έχουν λοιπόν να παίξουν και οι άνδρες ρόλο. Και το GAP 2, το σχέδιο δράσης 2, σίγουρα το λαμβάνει αυτό υπόψη. Δεύτερον, νομίζω ότι καθορίζει τους στόχους και ενώνει τις κουκίδες, να το πω έτσι. δηλαδή, ε, βλέπουμε πώς ε, ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξωτερικές της δράσεις ε, και έτσι συνδέουμε τις δράσεις ανάμεσα στην ΔΕΦΚΟ και άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και καθορίζουμε θεματικούς πυλώνες ε, την ε, καταπολέμηση της βίας εις βάρος ε, των γυναικών, την οικονομική ανδυνάμωση και κατόπιν έχουμε και την αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας. Έχουμε δει πρόοδο στην, στα παραδείγματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την δέσμευσή της για τη διασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων. Ε, από την Επίτροπο Νίμιτσα και ε, την υπατή ε, εκπρόσωπο Μογκερίνη. Είδαμε σημαντικές δράσεις και στην ΤΕΦΚΟ και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είδαμε σημαντικές δράσεις και στις αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης είδαμε πρόοδο καθώς και συνέργειες με τα ε, σημεία επαφής που δημιουργήθηκαν ε, για την ισότητα των δύο φύλων. Επίσης, επικεντρωνόμαστε στην ε, αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας. Μάλλον εδώ έχουμε και την περισσότερη πρόοδο. Φαίνεται ότι το σχέδιο Ράσης ΓΑΠ 2 έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τομέα αυτών, κυρίως επειδή περιλαμβάνει και κατάρτιση σε θέματα των δύο φύλων και είδαμε κάτι τέτοιο και σε αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κράτη-μέλη και ε, επίσης σε διάφορες ε, γενικές διευθύνσεις και συχνά η κατάρτιση αυτή προχωράει πέρα από απλά τη δημιουργία σημείων επαφής για την ισότητα των δύο φύλων πρόοδο είδαμε και στην συνεργασία. Είδαμε πολύ περισσότερο συντονισμό ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και τις ε, αποστολές, καθώς και ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη. Σε επίπεδο αποστολών είδαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στον εντοπισμό θεματικών στόχων και την εκπόνηση των εκθέσεων. Συνεχής παρακολούθηση των ε, σχετικών δραστηριοτήτων ε, είναι επίσης ένας από τους τομείς όπου είδαμε αρκετή πρόοδο. Σε αντίθεση με τον ΚΑΠ 1, όπου η παρακολούθηση ήταν περισσότερο ποιοτική φύσης και εθελοντική, στο σχέδιο δράσης ΚΑΠ 2 είναι υποχρεωτική σε αιτήσια βάση και βασίζεται σε αναλύσεις ε, όλων των αποστολών ε, καθώς και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο δράσης ΚΑΠ2 επίσης εξετάζει ποιες ε, αντιπροσωπείες σημειώνουν πρόοδο και ποιες όχι. Και στην έκθεση μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε Ε, σε ποιους τομείς ε, έχει ενσωματωθεί στις διάφορες δραστηριότητες ε, η πτυχή της ισότητας των δύο φύλων και που όχι. Επίσης υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές για την εφαρμογή σχετικών δραστηριοτήτων. άλλη έγγραφο με κατευθυντήριε γραμμέ που εστάλησε τι τις τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, φαίνεται όμω να αφορά κυρίω κυρίως δραστηριότητε τη ΤΕΦΚΟ. Επίση έχουν ε, αναλυφθεί δράσει ε, στο πλαίσιο του ΓΑΠ2. Έχουμε τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Οργανώνονται συναντήσεις με εταίρους μας για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της διαδικασίας παρακολούθησης, ε, συνεργαζόμαστε και με μη κυβερνητικέ οργανώσει. Δεν λαμβάνουμε δηλαδή αποκλειστικά πληροφορίε από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τα θεσμικά όργανα. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο στις Βρυξέλλες. Τέλος, ε, η διαθέσιμη χρηματοδότηση έχει βελτιωθεί. 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε συγκεκριμένα μέτρα. Και κατά την εξέταση των στατιστικών, ε, στην ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, βλέπουμε ότι σχεδόν το 60% των δραστηριοτήτων και της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΤΕΦΚΟ και της ΕΝΙΑ ε, στοχεύουν ε, στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα Έχουμε και την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών για τα δύο φύλλα. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Νομίζω λοιπόν ότι το βασικό μας μήνυμα όσον αφορά τα επιτεύγματα είναι ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει δέσμευση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να εξάγουμε σαφή συμπεράσματα σχετικά με το αν είναι σταθερή αυτή η πρόοδος και διαρκείας. Τέλος, ε, έχω εντοπίσει και κάποιες ελλείψεις. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Μιλώντας με διαφόρους, είχα την εντύπωση ότι ε, στην ΤΕΦΚΟ είναι πολύ πιο προηγμένη σε σχέση με αυτά που γίνονται στην ΕΙΕΔ. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, γυναίκες σε ε, ευάλωτη ε, θέση, καθώς και στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και τη διαμεσολάβηση. Μπορεί αυτή η εντύπωση να οφείλεται στο ότι πολλές πληροφορίες στην ΕΙΕΔΗ είναι εμπιστευτικές. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να έχουμε σαφή εικόνα του τι γίνεται εκεί. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΕΔ ομολογούν ότι πολλές πληροφορίες ε, είναι εμπιστευτικές και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να εξάγει κανείς συμπεράσματα. Δεύτερο θέμα είναι η έλλειψη σχέσης, ε, είναι ο, ο, ο κρίκος που λείπει ανάμεσα ο συνδετικός κρίκος που λείπει ανάμεσα στο εμπόριο και την ισότητα των δύο φύλων. Ε, ε, αν εξετάσουμε τις γενικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο, δεν ε, αναφέρονται οι γυναίκες. Το εμπόριο επηρεάζει και τις γυναίκες σε πολύ μεγάλο βαθμό και θετικά και αρνητικά. Και όταν έχουμε αυτή τη στρατηγική που υποτίθεται ότι είναι μια ενιαία θηρίδα για το θέμα αυτό, είναι κρίμα που δεν συμπεριλαμβάνεται και αυτό το θέμα. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως σε, σε ποσοτικά στοιχεία και όχι ποιοτικά. Η έκθεση παρακολούθησης δίνει πολλά αναλυτικά δεδομένα που δείχνουν πώς έχει σημειωθεί πρόοδος. Δεν γνωρίζουμε όμως Πώς επηρεάζουν τα προγράμματα αυτά τις κοινότητες υποδοχής, εάν οι δραστηριότητες που επιλέγησαν ήταν οι πιο κατάλληλες και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στις χώρες αυτές. Επίσης, σε πιο δύσκολες καταστάσεις, όταν έχουμε ευάλωτα κράτη ή ε, περιοχές σύγκρουσης, όπου υπάρχουν διάφοροι στόχοι στις, ε, για τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται, φαίνεται ότι το θέμα της ισότητας των δύο φύλων ε, γενικά τίθεται κατά μέρος. Και τέλος, πολλές από τις δραστηριότητες ε, στο πλαίσιο αυτό φαίνεται να είναι πολύ ευρείες και δεν είναι πολύ σαφές το πώς θα επιφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα με την εφαρμογή τους. Τι πιθανά ανοίγματα για το μέλλον υπάρχουν λοιπόν και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση και να ενσωματώσουμε καλύτερα την πτυχή της ισότητας των δύο φύλων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά ακούμε την προσέγγιση, την ολιστική προσέγγιση που ανακαλύπτει το σύνολο της κοινωνίας. Ε, να υπάρχει δηλαδή διασύνδεση ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές σε κυβερνητικό επίπεδο. Κάτι παρόμοιο μπορεί να γίνει σε επίπεδο κοινωνίας. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να συνεργάζονται με επιχειρήσεις και με άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό ομολογουμένως δεν είναι εύκολο σε ένα περιβάλλον όπου ε, ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών συρρυκνώνεται, αλλά οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι εάν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, νιώθουν λιγότερο απομονωμένες ε, στην χώρα τους, θα προστατεύονται και καλύτερα από το καθεστώς, από τις διάφορες συνομιλίες που είχα με μέλη της κοινωνίας των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια, για παράδειγμα. που δεν είναι αυτή τη στιγμή και το πιο δύσκολο περιβάλλον. Ε, ε, μου είπαν επανειλημμένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει τη σχέση με τις κυβερνήσεις. Δεν αρκεί η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, χρειάζεται περισσότερη πολιτική δέσμευση. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παίξει πιο σημαντικό ρόλο. Το διάγραμμα αυτό προέρχεται από μία έκθεση που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο McKinsey πρόσφατα το 2015 όπου ισχυρίζονται και προσπαθούν να δείξουν ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών. Μακροπρόθεσμα, ο ιδιωτικός τομέας θα υποφεληθεί αν επικεντρωθεί στις τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που ε, δημιουργούνται όταν βελτιωθεί η ισότητα των δύο φύλων. Και βλέπετε εδώ στο διάγραμμα ότι Μέχρι το 2025 θα μπορούσε να αναπτυχθεί πλήρως ε, το ε, ΑΕΠ παγκοσμίως ε, κατά 28 τρισεκατομμύρια δολάρια εάν διπλασιαστεί η συμμετοχή των γυναικών. Διατηρώντας σε σταθερό επίπεδο τη συμμετοχή των ανδρών. Αυτό είναι πολύ φιλόδοξο σχέδιο. άλλες ευκαιρίες για δράση. Συμπεριλαμβάνουν την ε, διασφάλιση ε, της μετατροπής σε πραγματική δράση της ε, πολιτικής δέσμευσης που ήδη υπάρχει, που μάλιστα υπάρχει σε πολύ ψηλά επίπεδα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΕΔ. Δηλαδή, η ισότητα των δύο φύλων να αποτελέσει προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα. Οι εμπειρογνώμονες λένε ότι σήμερα βλέπουμε κυρίως μια κατάσταση όπου οι πολιτικές αυτές είναι πιο πολύ τυπικής φύσης, ενώ όταν εφαρμόζονται ε, επικεντρώνονται κυρίως σε βασικά θέματα όπως είναι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η υγεία των μητέρων. Ε, ενώ θέματα όπως οι μεταφορές ή η γεωργία ε, θεωρούνται γενικά ουδέτερη, ε, ουδέτερη τομή ως προς το γένος, ενώ δεν είναι. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη απλούστευση της παρακολούθησης, το οποίο σημαίνει ότι Αυτή τη στιγμή η ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων ε, επισυνάπτεται σε πολλά έγγραφα αντί να ενσωματώνεται σε αυτά. Επίσης, πολλές μελέτες ε, δεν προχωρούν αρκετά εις βάθος ώστε να βοηθήσουν ε, στην εκπόνηση εγγράφων δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το ομολογεί και η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΙΕΔ υπάρχει ανάγκη. Η ισότητα των δύο φύλων αναφέρεται στις ε, εμπορικές διαπραγματεύσεις ε, και την παρακολούθηση των εμπορικών ε, συμφωνιών. Πολλοί εμπειρογνώμονες μιλάνε για καλύτερη τεκμηρίωση της δυναμικής των δύο φύλων στην παροχή υπηρεσιών, στη δημιουργία προτύπων και στους κανονισμούς και να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη το θέμα των δύο φύλων και στις μελέτες αντικτύπου. Άλλοι επιρογνώμονες ε, μιλούν για ε, την ε, ενσωμάτωση σε εμπορικές συμφωνίες των εργασιακών δικαιωμάτων. Επίσης, θα πρέπει οι άντρες να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των δύο φύλων. Θα πρέπει δηλαδή να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των ε, ανδρών και αυτό ε, φαίνεται από την έκθεση της ΕΕ. Επίσης, θα πρέπει να ε, έχουμε καλύτερη προσαρμογή στην τοπική πραγματικότητα. Διάφορες δημογραφικές, οικονομικές, διάφοροι δημογραφικοί και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την κατάσταση των γυναικών και πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ε, στις διάφορες χώρες. Μπορεί γενικά να φαίνεται ότι είναι παρόμοια, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζετε ότι κάθε περιφέρεια, κάθε χώρα έχει ιδιαίτερες ε, ε, παραδοσιακές δομές και γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμόσουμε καλύτερα τις δράσεις μας στα μέτρα ε, των διαφόρων χωρών. Θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τον ρόλο των ε, αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν, μπορούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στις επαφές με κυβερνήσεις και τοπικούς παράγοντες, να ε, συντονίζουν τις δράσεις ε, των κρατών μελών ε, στη χώρα και να είναι και ένα πρώτο σημείο επαφής για τους διεθνείς εταίρους. Χρειάζονται όμως περισσότερους ανθρώπινους πόρους. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζουμε τις γυναίκες ως παράγοντες, όχι ως θύματα. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε το ρόλο των γυναικών ε, στην ε, δικαιοσύνη, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους ε, στην δημόσια ζωή και στις έρευνες. Και δύο τελευταία που θέλω ακόμα να αναφέρω. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση που θα μπορούσε να παρέχεται όχι μόνο σε αυτούς που ασχολούνται με τα θέματα αισιότητας των φύλων, αλλά και στην ενδιάμεση ιεραρχία της Επιτροπής των Αντιπροσωπιών και να διατίθεται τέτοια κατάρτιση και σε μη καπόμικρον και άλλους φορείς στην κάθε χώρα όπως και να δεσμευόμαστε μακροπρόθεσμα και η ΕΔ το υπογραμμίζει το θέμα αυτό δηλαδή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειες αυτές θα έχουν καρπούς, χρειάζεται να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και σαφή χρονοδιαγράμματα. Ε, συνολικά θα έλεγα ότι το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε μία ισορροπημένη υγιή βάση ώστε να θεωρήσουμε ότι έχει ενσωματωθεί απολύτως η διάσταση του φύλου στην διάσταση της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν με σωστό τρόπο ώστε να έχουμε και σωστά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος, την κυρία Ιωαννίδη για την παρουσίαση της μελέτης αυτής και θα ήθελα τώρα να ρωτήσω αν τα μέλη έχουν κάποια ερώτηση ή παρατήρηση για την μελέτη αυτή. Αν όχι, θα πάμε στο επόμενο σημείο της ημεσίας διατάξεως, την υλοποίηση του κοινού εγγράφου εργασίας για την ισότητα των φύλων και την ε, προσαρμογή των, ε, της ζωής νεαρών κοριτσιών και γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων. Η κυρία Μακάβαν και η κυρία Σούιτσα ε, έχουν, είναι, έχουν εργαστεί εδώ και θα τους δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την διοργάνωση αυτής της κοινή συνεδρίας μεταξύ των δύο επιτροπών μας. Ευχαριστώ την κυρία Ιωαννίδη που μας έδωσε ένα πλαίσιο για την γνωμοδότησή μας. Ε, η κυρία Σούικα δεν μπορούσε να είναι εδώ άμεσα και την εκπροσωπώ εγώ προς το παρόν. Εδώ έχουμε μια έκθεση λοιπόν εφαρμογής, υλοποίηση. Εδώ δεν συζητούμε κατά πόσον θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο δράσεως για την ισότητα των φύλων. Αυτά τα είχαμε συζητήσει πέρυσι για το περιεχόμενο κτλ. Τώρα πρέπει να δούμε κατά πόσον λειτουργεί, κατά πόσον προχωρεί προς την σωστή κατεύθυνση και κατά πόσον πρέπει να το προσαρμόσουμε. Ήθελα λοιπόν απλώς να θυμίσω στα μέλη γιατί έχουμε ένα νέο πρόγραμμα. Το προηγούμενο ήταν πολύ στενό, αφορούσε μόνο την γάμα δελτα και όχι την, το σύνολο της εξωτερικής διάστασης. Και είχαμε μία περισσότερο άσκηση επιλογής πεδίων με τσεκάρισμα. Οι αντιπροσωπείες ε, συνήθως ανέθεταν στο νεότερο μέλος, συνήθως γυναίκα, της αντιπροσωπείας τη σχετική αυτή δουλειά, τσεκάραμε τα παιδεία που έπρεπε και το αποστέλαμε στις Βρυξέλλες. Δεν ήταν μια πολύ πλήρης προσέγγιση. Στον πολιτικό μας διάλογο δεν ετέθη ποτέ το θέμα. Δεν ήταν κάτι με το οποίο ασχολούνταν, αν θέλετε, οι πιο ισχυροί, οι πιο σοβαροί συνάδελφοι. Ενώ στο νέο πρόγραμμα έχουμε τρεις θεματικούς πυλώνες για ψυχολογική ισορροπία, για την προαγωγή οικονομικών δικαιωμάτων και την ενίσχυση των φωνών τους και τη συμμετοχικότητός τους. Αλλά με μεγάλη έμφαση στην θεσμική αλλαγή που θα πρέπει να γίνει ώστε ο μηχανισμός συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνει υπόψη του το θέμα αυτό οι σημαντικέ αλλαγές και πολιτισμικά που έχουν γίνει είναι ότι πλέον το θέμα δεν αντίθεται σε κάποιο νέο μέλος αντιπροσωπεία, αλλά είναι καθήκον του επικεφαλής. Και το 85% των αντιπροσωπείων έχουν πλέον υποβάλει τι αναφορές τους για τους πόρους που έχουν καταναμηθεί, για τις αναλύσεις ισότητα των φύλων επί τη βάση της χώρας που έχουν γίνει. Δεν ξέρω πόσες τέτοιε έχουμε δει. Θα έπρεπε να τι ζητούμε για κάθε χώρα για να μπορούμε να υποβάλουμε ερωτήσει. Γιατί αυτές τι αναλύσεις όταν, όταν εξετάζουμε τα σχετικά θέματα στι επιτροπές δεν τι έχουμε. Για να ξέρουμε και τι ρωτούμε. Ελάχιστα πρότυπα για το gender mainstreaming, καταμέτρηση, ποσοτικοποίηση πόσες από τις μελέτες και εκθέσεις μας ασχολούνται με το θέμα αυτό. Κατά μέτρηση των αποτελεσμάτων, δηλαδή όταν προσμετρούμε την επιτυχία των προγραμμάτων, πόσα από αυτά ήταν επωφελή για τις γυναίκες. Εδώ λοιπόν δεν θέλω να επαναλάβω γιατί, τα γιατί, τις αιτίες του προγράμματος, αλλά την κατεύθυνση και την επιτυχία του. Εμείς συναντήσαμε κάποιους από τους ε, πρέσβεις μαζί με την κυρία Σούικα. Οι πρέσβει έρχονται στις Βρυξέλλες πλέον ε, μία φορά το χρόνο για να συναντηθούν με τους προσώπους της ΕΔ και της Επιτροπή και νομίζω ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να τους τίθενται από τους Επιτρόπους. Εν πάση συναντήσαμε Κάποιου πρέσβει. είχαμε δύο ακροάσεις και διαρρήσαμε τι συστάσεις σε κατηγορίε. Μία για την Επιτροπή και την ΙΕΔ αν θέλετε δηλαδή για, το, για την κεντρική δομή της διοίκηση. δεύτερον για τι αντιπροσωπείε. και τρίτον συστάσεις για το ίδιο το Κοινοβούλιο. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομίζω ότι οι σχετικέ δράσει πηγαίνουν προ την κατεύθυνση. Βλέπω και την Γαμαδέλτα Ντεύκο, τον Ζανλουί Βιλέ που έχει κάνει πολλή δουλειά εδώ. Αλλά πρέπει να δούμε και τι υπόλοιπε εξωτερικέ γενικέ διευθύνσει. Δεν είναι μόνο η Ντεύκο. Είναι και θέμα τη ΝΙΑΡ, e τη Trade, τη ΙΕΔ. E Χρειαζόμαστε μια οριζόντια προσπάθεια και πρέπει να μα πούνε ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά τα θέματα για να υπάρξει συντονισμός και να γνωρίζουμε περισσότερα. Ακούσαμε και δηλώσεις επιτρόπων ότι θα εστιαστούν στα θέματα αυτά και θα τα προωθήσουν ζωηρά. Αλλά πρέπει να ακούσουμε και περισσότερα. Ακούσαμε για τα κενά στην ε, εμπορική πολιτική, αυτό είναι σωστό. Εγώ ήμουν πρόσφατα στο Μπαγκλαντές, στο οποίο υπάρχει ένα δυνητικό πρόβλημα ακριβώς για τον σεβασμό των προτύπων ILO, το οποίο σχετίζεται σε πολύ σημαντικό ποσοστό με τις γυναίκες. Με τις γυναίκες που έχουν καταστεί η βασική, το κυρίαρχο εισόδημα για την οικογένειά τους, για τον οικοκυριό τους, μεταξύ άλλων. Πρέπει λοιπόν να δούμε και το θέμα των γενικών ως βασικών φορέων, παικτών στο παιχνίδι και όχι μόνο ως δεκτών. Πέρυσι ήμουν στην Κένια και συναντήθηκα με κάποιες ε, γυναίκες στις τοπικές κυβερνήσεις και με ρωτούσαν οι καταπληκτικές αυτές γυναίκες ε, τι συμβουλές μπορείτε να μας δώσετε. Ε, γιατί κινούνται, γίνονται πολλά πράγματα σε διάφορες χώρες. Αλλαγή λοιπόν στην κεντρική διοίκηση. Στι αντιπροσωπείε βελτιώνει το πράγμα. Το 85% όπω σα είπα έχουν υποβάλει έκθεση για την ισότητα φύλων και το 58% των νέων έργων έχουν διάσταση φύλου. Και οι αντιπροσωπείε μας ζήτησαν προτεραιότητες για να εστιαστούν υπό κάθε έναν από τους πυλώνε. Αυτό είναι καλό ως εκκίνηση, αλλά με κατά πόσον θα έπρεπε να επιλέγουν περισσότερα από, περισσότερες από μία θεματικές, γιατί είχαμε την προτεραιότητα από την Επιτροπή της Βίας κατά των γυναικών, αλλά δεν θέλουμε να τις βλέπουμε μόνο ως θύματα, θέλουμε να τις βλέπουμε ως ηγέτιδες. Σε θέματα των μεταφορών, της υγείας, πριν γίνω μέλος του Κοινοβουλίου, ασχολούμεν με την τοπική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο και όταν είχαμε ζητήσει για το πώς θα πρέπει να σχεδέσουμε αισθήματα μεταφορών ενός γυναικών είχαν πολύ διαφορετικέ απαντήσεις από, ότι, από τους άνδρες. Επομένως πρέπει να δούμε ευρύτερα τα θέματα. Γνωρίζουμε ότι και στα τραπεζικά και τα χρηματοπιστωτικά πρέπει να έχουμε, να ρωτούμε τη γνώμη των γυναικών. Η ανάλυση φύλου έχουμε σημαντικό κενό από τις χώρες και τις σχετικές αναλύσεις. Πρέπει να ακούσουμε από την Επιτροπή βεβαιώσεις ότι οι αναλύσεις αυτές γίνονται και ότι τις λαμβάνετε. Και είναι ένα δυναμικό έγγραφο ή είναι απλώς άσκηση να τσεκάρουμε τα κουτάκια που έλεγα πριν. Και οι αναλύσει αυτέ πρέπει να γίνονται με, σε συνδυασμό, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ενώσει. Δεν είναι απλώς τι θα λέει η κάθε κυβέρνηση, θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη ματιά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και κάποιες ε, συστάσεις για εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Γιατί και εμεί, όταν συναντόμαστε με τους επικεφαλείς αντιπροσωπείων πρέπει να θέτουμε τα θέματα αυτά. Εγώ συνάντησα μία συνάδελφο που ήταν στην ΟΑΣ την προηγούμενη εβδομάδα και ρώτησε σε διάφορες συνεδριάσεις για τα θέματα των γυναικών και οι άλλοι ε, γούρλαν τα μάτια τους. Δεν γίνεται να μην έχουμε συνεχή ενημέρωση για το θέμα αυτό. Ίσως θα πρέπει να έχουμε και μια αιτήσια συζήτηση για το θέμα αυτό και να υποβάλουμε έκθεση κάθε τρία-πέντε χρόνια για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η Επιτροπή Γυναικών νομίζω θα πρέπει να το λάβει υπόψη της αυτό. Και άλλο ένα στοιχείο που είναι περισσότερο για την Κομισιόν. Δεν έχουμε τους ίδιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Μάλλον πώς σχετίζονται όλα αυτά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την επίτευξή τους. Και καθότι άκουσα και τους προηγούμενους ομιλητές, ε, σκεπτόμουν ότι μία από τις σε ένα πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων πρέπει να αφορά και στα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχουν διάφορα διμερή έργα και προγράμματα και ίσως θα πρέπει να έχουμε μία σύσταση και για τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρξει πιο ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Σε ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ την συνεισηγήτρια. Θα δώσω τώρα. Θα ήθελα μάλλον να δώσω το λόγο στη άλλη συνεισηγήτρια την κυρία Σούσα που δεν είναι όμως εδώ από την δικιά μας επιτροπή. Η κυρία Κοσλόφσκα όμως την αντικαθιστά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τη Λίντα Μακάβιν. Πολλά είπε, είναι σημαντικά συμφωνώ με κάθε πρότασή της. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση αυτή. Και το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν για την απουσία της κυρίας Σούκα που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, όμως έγραψε κάποια πράγματα τα οποία και θα σας διαβάσω. Μου ζήτησε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσοι δούλεψαν για αυτή την υπόθεση. Όπως ξέρετε, η αρχή ισότητας ανδρών γυναικών έτσι κι αλλιώς εγγραφέται στις συνθήκες και συνεπώς πρέπει να προωθείται σε όλες τις δραστηριότητε, σε όλα τα μελλοντικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα συνολικής ε, δράσης αναφέρεται σε αρχές για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, σε φιλοδοξίες επίσης για την ισότητα αυτή. Τώρα, με αυτή την έκθεση εφαρμογής θέλουμε να επικεντρωθούμε με την κυρία Μακάβιν στα αποτελέσματα και στις συστάσεις για το μέλλον. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε έχοντας υπόψη μας ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τον ΚΑΠ 2 και έχουν σημειωθεί θετικές στάσεις. Αυτό που επίσης θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, γίνονται επικοδομητικές ε, προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία επίσης με την κοινωνία των πολιτών, ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, ανάπτυξη online αναφορά σε περίπτωση που υπάρχουν παραβιάσεις για να ενημερώνονται τα όργανα. Θέλουμε επίσης να υπογραμμίσουμε ότι προσβλέπουμε στις προτάσεις σας, στις απόψεις σας και η κυρία Σούκα πιστεύει ότι η σημερινή συνάντηση θα συνεισφέρει ε, προς αυτόν τον σκοπό και προς την ισότητα των δύο φίλων. Και τώρα θέλω να προσθέσω και λίγα πράγματα εκ μέρους μου. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι η αλλαγή γλώσσας και νοοτροπίας είναι κάτι αναγκαίο. Το να αρχίσουμε να μιλάμε για τις γυναίκες ε, όχι ως θύματα, αλλά ως ε, εκείνες που έχουν τα πράγματα στα χέρια τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η γλώσσα μας μερικές φορές δεν είναι κατανοητή από τις γυναίκες που βρίσκονται σε αυτή τη δυσάρεστη θέση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε πράγματα τα οποία να είναι πραγματικά και πολύ σημαντικά για αυτές και τις οικογένειές τους. Όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των ε, γυναικών εργαζομένων, είναι πολύ βασικό. Οι γυναίκες είναι θύματα καταχρήσω πολλές φορές οικονομικά, εκμετάλλευσης, Οπότε αν τις βοηθήσουμε να αγωνιστούν για τα εργασιακά τους δικαιώματα, είναι κάτι το οποίο μπορούν να αντιληφθούν. Και το να μιλάμε γενικά για την εφαρμογή είναι ζωτική σημασία. Γιατί μιλάμε για δικαιώματα παντού και γίνονται πάρα πολλές κενές περιεχομένου δηλώσεις. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι στο χαρτί σύμφωνοι, αλλά ακόμα πιο δύσκολο είναι να γίνει και κάτι στην πράξη. Συνεπώς η εφαρμογή αυτή είναι πολύ σημαντικό πράγμα για το θέμα μας. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και τις δύο εισηγήτριες και προσθέτω ότι ο τρόπος που συνεργάζεστε με συναντήσεις, με πρέσβεις είναι κάτι το οποίο εκτιμούμε όλους ιδιαίτερως. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, Λί Πρόεδρος. Και τώρα, η Σκιώδης, πρώτα απ' όλα, κύριος Μαρσελίση. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι διπλά σκιώδης εισηγητής, γιατί είμαι στην Τέδα, αλλά μιλάω και εκ μέρου του κύριου Σόλε που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, που είναι από την Επιτροπή Γυναικών. Λοιπόν, συμφωνούμε και χαιρόμαστε για τις βελτιώσεις που έχουν γίνει ανάμεσα στο GAP 1 και το GAP 2. Έχουν γίνει ουσιαστικές βελτιώσεις για τις οποίες πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας. Ε, συγχρόνως όμως δεν πρέπει να είμαστε τόσο θετικοί γιατί πολλοί δρόμος μένει ακόμα να διανύσουμε. Πολλά μένουν να γίνουν για να φτάσουμε στους gender champions που υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες που ακόμα δεν έχουν καν ε, θέσει σε ισχύ το δικό τους πρόγραμμα δράσης. Οπότε να το επενθυμίζουμε και αυτό. Συμφωνούμε επίσης με τις συνεισηγήτριες. Όντως πρέπει να διευκολύνονται οι επικοινωνία, η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, αλλά πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι δυστυχώς τα θέματα του φύλου δυστυχώς αποσιάζουν από τους πολιτικούς διαλόγους, από τις αξιολογήσεις, δεν θεωρούνται κύρια ζητήματα, προτεραιότητα, όχι, είναι εκτός των ε, αποφάσεων. Μ' άρεσε αυτό που είπε και η συγκέντρια πριν για το εμπόριο και το φύλλο. Όντω δεν υπάρχουν πολλά πράγματα γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εμπορικέ συναλλαγές με χώρε όπου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, συμβαίνουν φοβερά πράγματα όπως το Μεξικό ε, που εξαφανίζονται γυναίκες. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό αυτό το missing link αυτό που ο κρίκος που λείπει δηλαδή να μπει. Να υπενθυμίσουμε επίσης και το ρόλο των γυναικών. Όντως, με το προσφυγικό είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες ήταν τα κύρια θύματα. Είναι εκείνε που υποφέρουν περισσότερο από όλη αυτή τη διαδικασία μετανάστευσης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι γυναίκες αυτές να έχουν κεντρικό ρόλο στον προβληματισμό μας. Να τονίσουμε λοιπόν επίσης όχι μόνο τα θετικά, τα επιτεύγματα δηλαδή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη Εξωτερική Δράση, αλλά να δούμε λίγο τι γίνεται και με κυρώσει σε χώρες ή σε αντιπροσωπείες της Κομισιόν όπου δεν γίνονται αυτά που θα πρέπει να γίνονται, που προβλέπουν τον ΚΑΠ 2, για παράδειγμα, οι στόχοι της χιλιετίας. Δεν έχω ολοκληρώσει, οπότε παρακαλώ λίγη ησυχία στην αίθουσα, λέει ο μιλητή. Τέλος υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το σχέδιο δράσης να προωθηθεί, πρέπει να βελτιώσουμε και την κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με αυτό το ζήτημα, αλλά χρειάζεται και περισσότερο προσωπικό ειδικευμένο στα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων γιατί δυστυχώ πρόκειται συνήθως για ανθρώπους που έχουν άλλε αρμοδιότητες, άλλη επιμόρφωση και αναλαμβάνουν το θέμα το, της ισότητας των δύο φύλων και άρα δεν του δίνουν την προτεραιότητα που θα έπρεπε. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε ότι μπορείτε να βασιστείτε και στον Ζόρτη και σε μένα για να προχωρήσουμε με την έκθεση αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Um, On behalf of my colleague... Uh, Μιλώ εκ μέρου τη συναδέλφου Ιλιάνα Ροντρίγε που ναι, ζητεί συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα ε, που δεν μπόρεσα να ακούσει την παρουσίαση της έκθεσης ε, και την ανταλλαγή απόψεων πάνω στο σχέδιο έκθεσης. Ε, διαβάζω λοιπόν τα λόγια τη. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές για τη δουλειά τους ε, που αποτελεί πολύ καλό σημείο κίνησης. Ε, βρισκόμαστε στο πρώτο έτος της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την ισότητα των δύο φύλων 2. Γι' αυτό είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε τι πάει καλά και τι πρέπει να βελτιωθεί, διότι έχουμε ακόμα χρόνο να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις. Έχουμε τους τρεις θεματικούς πυλώνες και τον οριζόντιο πυλώνα και σίγουρα αποτελούν πολύ θετικές πτυχές. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει εάν δεν αλλάξουμε την ε, θεσμική νοοτροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα ήθελα και εδώ να προσθέσω ε, τη δική μου προσωπική παρατήρηση ότι είμαι πολύ περήφανη που ήμουν ισκιώδης συγγήτρια για την έκθεση για την ισότητα των δύο φύλων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και ορατή δουλειά. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί θετικά στοιχεία στον πυλώνα αυτών για την ενδυνάμωση των γυναικών ε, και ε, στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αυτά όμως δεν ακούν, Όπως μας δείχνει η μελέτη του EPRS, το GAP 2 Ε, επικεντρώνεται δυσανάλογα στα ποσοτικά δεδομένα και αναλύσεις. Ε, μας λείπουν όμως ποιοτικά δεδομένα που θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε σωστά τα αποτελέσματα των δράσεων ε, καθώς και τα ωφέλη και τους κινδύνους τους. Υπόθηκε ήδη σήμερα ότι δίνουμε προτεραιότητα στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Θα πρέπει όμως να επιφέρουμε ποιοτικές αλλαγές διαρκείας και η ευρεία φύση πολλών από τις δραστηριότητες ε, ε, καθιστούν πολύ δύσκολη την ε, διαπίστωση πρόοδου. Αυτή την εβδομάδα πήγα στην Πορτογαλία με αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΦΕΜ και σε αυτή την αποστολή και σε πολλές άλλες διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι δήμοι και οι περισσότερες κυβερνήσεις των κρατών μελών ε, έχουν φιλόδοξα σχέδια για την ισότητα των δύο φύλων. Αυτό που συχνά λείπει όμως είναι η αξιολόγηση των δράσεων που εφαρμόζεται και αυτό είναι πρόβλημα και εδώ. Βέβαια, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι εφαρμόζονται οι προτινόμενες δράσεις. Είναι όμως ακόμη πιο σημαντικό να γνωρίζουμε εάν επιφέρουν τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Εάν δηλαδή πηγαίνουμε προς την κατάλληλη κατεύθυνση ή αν θα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Και να μην ξεχνάμε ότι οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ε, και τις ε, διάφορες ε, συνθήκες και τις διάφορες προτεραιότητες των διαφορών κρατών και περιφερειών. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ακριβή δεδομένα και πριν και μετά την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς το μέτρο Χ έχει καταφέρει να μειώσει την, τον γενετήσιο ακροτηριασμό των γυναικών σε μια περιφέρεια ή την βία βάρους των γυναικών σε άλλες περιοχές και με τι ποσοστά. Τι δεν λειτουργήσε καλά. Πρέπει να απαιτήσουμε τέτοιου είδους δεδομένα. Δεν είναι σαφές αν ε, τα δεδομένα ε, που έχουν επιλεγεί ήταν τα πιο κατάλληλα. Συχνά ε, αυτά εξετάζονται με πολύ γενικό και αφηρημένο τρόπο και αυτό ακριβώς θα πρέπει να αποφύγουμε. Θα πρέπει να ενεργήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο σε τοπικό επίπεδο και σύμφωνα με την έκθεση για το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα ε, βλέπουμε ότι ε, από τότε που ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων το 2006 έχουμε αύξηση του χάσματος και Σύμφωνα με τα δεδομένα, αυτή τη στιγμή θα απαιτήσει 100 χρόνια για να κλείσει το χάσμα σε σχέση με 83 χρόνια πριν 12 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν πολύ γρήγορα να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις. Ε, είναι χρήσιμα τα μέτρα εάν επιφέρουν πραγματικές απτές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Ε, δεν αρκούν τα λόγια στο χαρτί, θα πρέπει αυτός να είναι ο στόχος μας, ε, αλλιώς δεν θα αξίζουν τον κόπο οι προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ward. Να στραφώ στους εκπροσώπους της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη. Φαντάζομαι ότι έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Κοιτάζω και το ρολόι. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, να ευχαριστήσω την κυρία Ιωαννίδη για την παρουσίαση και την μελέτη και πάω απευθείας στο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες, δεν έχουμε πάρα πολλά υποχρεωτικά μέτρα. Μας έλειπαν 22 από τις συνολικές ε, εκθέσεις των αντιπροσωπιών Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Γενέβη είναι πιο εύκολα εξηγήσιμε. αλλά θα προσπαθήσουμε, θα συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας να φτάσουμε στο 100% του χρόνου. Μας λείπουν όμως και σημαντικά πεδία όπως εκείνο της ΓΔ Trade, το οποίο ετέθηκε στην έκθεση και επί της ουσίας. Έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας και έχουμε δεσμευτεί όχι να βρούμε λύσει γιατί δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε κάτι από όλα αυτά, αλλά έχουμε δεσμευτεί να υποβάλουμε πληρέστερες και τακτικότερε εκθέσεις. Για τις εκθέσεις των κρατών μελών ε, ασκούμε πίεση. Ήμουν στο Συμβούλιο πριν έρθω εδώ και όλους τους πιέζουμε να υποβάλουν τι σχετικέ εκθέσει. Τώρα, τα το θέμα του εμπορίου. αναφέρεται στις μελέτες ότι είναι ένα μέσο που θέλουμε να διαρευνήσουμε και να εξετάσουμε από κοινού με τη γάμα δέλτα γιατί δεν το έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Γιατί εδώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η διάσταση του φύλου θα λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές. Υπάρχουν άλλες περιοχές, για παράδειγμα, όπου έχουμε καταβάλει προσπάθειες να είμαστε πιο ποιοτικοί και λιγότερο ποσοτική. Για το θέμα της ποιότητας έχετε δίκαιο και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά για να έχουμε ποιότητα πρέπει να έχουμε πρώτα ποσότητα, λέει ο μιλητής, δηλαδή δεδομένα. Δεδομένα για το διαχωρισμό των φύλων, χωρίς τα οποία δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου ενός έργου, ενός προγράμματος, ενός μέτρου για το γενική πληθυσμό συνολικά. η σύγκριση ποιοτικών αξιολογήσεων ε, που προέρχεται από την Ζάμπια ή την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έτσι επί παραδείγματι μπορεί να μην είναι συγκρίσιμη με μια άλλη. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικώς συγκρίσιμα στοιχεία και όχι να συγκρίνουμε μήλα με αχλάδια. η υποβολή εκθέσεων είναι σημαντική. Αναφερθήκατε στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο που έχουμε θεσπίσει, ώστε να ευθυγραμμιζόμαστε με τους στόχους και να έχουμε μία ενιαία υποβολή εκθεσής που να μας δίνει μία δίκαιη, πλήρη δηλαδή εικόνα για το πώς θα πηγαίνουμε. Πώς καλύπτουμε το κενό για τους στόχους αυτούς SDG. Που είναι οι στόχοι προς, τους, την κατεύθυνση των οποίων εργαζόμαστε όλοι. Τώρα πολλά ακόμα θα μπορούσε να πει κανείς αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω. Γιατί όπως γνωρίζετε θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες για το ζήτημα αυτό. Αλλά θα σταματήσω αυτό και με χαρά να συμμετάσχω σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις σας επί του θέματος. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εσάς και να ενημερώσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 14 Νοεμβρίου 5 το απόγευμα. Η επόμενη κοινή μας συνεδρίαση είναι 4 Δεκεμβρίου για την εξέταση τροπολογιών ακριβώς. Ευχαριστώ λοιπόν την ε, συμπρόεδρο, ευχαριστώ όλα τα μέλη και θα, ξεκινη... θα συνεχίσουμε τώρα με τα θέματα της Επιτροπής Γυναικών. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.